Okay, colleagues, if everybody is back... Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα που γύρισαν όλοι στην αίθουσα και όλες, βλέπω ότι και ο κύριος Ρόμεβα έχει βάλει το κατάλληλο μπλουζάκι για το επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Είναι ένα μπλουζάκι που γράφει άκτον άκτα. Έχουμε λίγα λεπτά καθυστέρηση. Um... The last week the uh, EDPS Λοιπόν, δεύτερη γνωμοδότηση για την άκτα και συνεχίζουμε. Θα ακούσουμε τον κύριο Μπουταρέλη του EDPS, αλλά όμως πριν από αυτό θα ζητήσω από τον εισηγητή να μας δώσει μία σύντομη επικαιροποίηση ε, για τα διαδικαστικά, ο κύριος Ρούτσας. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, ε, κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι συζητούμε το θέμα αυτό, συζητεί το θέμα αυτό επί της ουσίας στην Ίντα. Ε, στην Ίντα λοιπόν το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ σφιχτό. Ζητήσαμε να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, ζητήσαμε την Ίντα να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε να ε, συζητήσουμε καλύτερα το θέμα, να το προετοιμάσουμε καλύτερα. Γι' αυτό η Ίντα δέχτηκε τελικά να μας δώσει μερικούς, μερικές εβδομάδες. Επομένως, χρονοδιάγραμμα είναι ως εξή. Παρουσίαση της, ε, του σχεδίου έκθεσης την 8η Μαΐου. Να σας πω ότι ε, η γνωμοδότηση ήδη, το προσχέδιο της ήταν έτοιμο περί την 3η Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και εμείς σε πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών θα είναι η 9η Μαΐου. Μη διαμαρτύρεστε, να τελειώσω. Έτσι ώστε να έχουμε όλες τις γλωσσικές εκδοχές των τροπολογιών ή, εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ναι, ε, ε, ε, ότι θα έχουμε σαν βάση σε το αγγλικό κείμενο, τότε η υποβολή θα μπορούσε να είναι 14, θα μπορούσε να είναι 14 Μαΐου. Κοιτάξτε, δεν τα αποφάσισα εγώ αυτά όλα μόνος μου. Σας είπα και προηγουμένως ότι εξαρτώμεθα από την ίντα. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η ίντα την τελευταία στιγμή πήρε την απόφαση να μην ε, προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να ε, επιλέξει γρήγορη διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προθεσμία που είχε ε, βάλει εξ αρχής η ΙΝΤΑ ήταν ακόμα σφιχτότερη. Τους Ελπίσαμε να το μεταθέσουν για μερικές εβδομάδες αλλά, ε, και το έπραξαν, αλλά δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει αρκετά σφιχτό το χρονοδιάγραμμα. Η ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή μας θα πρέπει να λάβει χώρα την 30-31η Μαΐου. We are also ε, planning of having a workshop for our, for, our, for, the Committee ε, between the ε, και μεταξύ 9ης και 15ης ε, Μαΐου η Γραμματεία θα είναι σε θέση να μας δώσει τις ακριβείς ημερομηνίε για, για το εργαστήριο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι αυτό το σφιχτόχρονο διάγραμμα όντω το καταλαβαίνω ότι δημιουργεί δυσκολίε. Δεν το αποφάσισα εγώ όμω και σίγουρα δεν ήταν ένα δικό μα θέμα. Ο κ. Μπουζούτιλ, διαδικαστικό. Ναι, δεν, δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι αυτό το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, μία μέρα περιθώριο για να υποβληθούν τροπολογίες ε, για μία γνωμοδότηση τόσο σημαντική που είναι γνωμοδότηση υπό το άρθρο 36 ε, από την 8η στην 9η Μαΐου, πραγματικά είναι υπερβολικά μικρό το χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να το ξανασχεδιάσουμε το χρονοδιάγραμμα. συμφωνήσαμε να ζητήσουμε περισσότερο χρόνο από την Ίντα. Μας δόθηκε ο χρόνος αυτός και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να δουλέψουμε έχοντας περισσότερο χρόνο για τις τροπολογίες, γιατί διαφορετικά στην ουσία θα μας ζητηθεί να ψηφίσουμε επί της ε, ε, απόψεως του συντάκτου, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα υποβολής τροπολογιών. Γι' αυτό ζητώ ε, αλλαγή του χρονοδιαγράμματος, έτσι ώστε τα μέλη να έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν την ησυχία του τροπολογίες. Προεδρό ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Όχι οι συντονιστές ε, να μιλήσουν ε, για να αποφανθούν επί των διαδικαστικών και μετά να πούμε ε, τι θα γίνει, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, 3η Μαΐου είπατε, όχι, όχι, δεν είπαμε αυτό, είπαμε ότι το προσχέδιο θα υποβληθεί επισήμως την 8η Μαΐου, αλλά θα είναι διαθέσιμο ήδη περί την 3η Μαΐου. Είναι και θέμα γλωσσών, εάν θα πρέπει να μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες, αν θα συμφωνήσουμε να δουλέψουμε μόνο με το αγγλικό έγγραφο, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της εργασίας μας. Και το ξαναλέω και το τονίζω, ούτε κι εγώ είμαι ευχαριστημένος. Προσπαθήσαμε να δούμε όλες τις δυνατότητες, πιθανότητες κτλ. Ε, ε, καταφέραμε να πείσουμε την Ίντα να μας δώσει αυτές τις μερικές εβδομάδες περιθώριο, αλλά ε, ζητώ την κατανόησή σας για μία ακόμα φορά. 3η Μαΐου θα έχετε διαθέσιμο το κείμενο στην Αγγλική. Αυτός είναι ο στόχος μας. Επίσημώ όμως θα υποβληθεί την 8η Μαΐου. Ε, θα δώσω το λόγο σε έναν συνάδελφο, συντονιστή των φιλελευθέρων και μετά, ε, μετά την παρέμβαση του κ. Μπουταρέλη θα ε, τους δώσω το λόγο. πριν ναι, Έχω μία απορία. Κανονικά, όταν πρόκειται για διεθνή συμφωνία και το Κοινοβούλιο απλώς γνωμοδοτεί ή έχει συμβουλευτικό ρόλο, η γνωμοδότηση είναι υπέρ ή κατά απλώς. Άφηστε με να ρωτήσω Δεσποινής. Λοιπόν, ο εισηγητής αυτό θα κάνει ή η γνωμοδότησή του θα έχει μήπως πολλές συστάσεις για να καταλάβουμε τι αφορούν οι τροπολογίες. Δεν καταθέτουμε τροπολογίες για το επεξηγηματικό σημείωμα. Κοιτάξτε, θα είναι μάλλον σαν ψήφισμα, όχι απλώς σύσταση ναι ή όχι. Γιατί είναι βάση του άρθρου 36 που απαιτεί από την Επιτροπή μας να γνωμοδοτήσει για τη συμβατότητα με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τώρα που το εξηγήσαμε αυτό, ό,τι άλλο θέλουμε να πούμε, να τα πούμε στους συντονιστάς. Έχετε διαδικαστικό κύριε Μπουζουτήλ. Ναι, διαδικαστικό. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στις 3 Μαΐου είναι την επόμενη εβδομάδα. και δεν μπορούμε να συναντηθούμε μέχρι τότε και στις 9 Μαΐου αν είναι σωστό το ημερολόγιό μου είναι αργία δεν μπορούμε στις αργίες να Πότε θα το συζητήσουμε λοιπόν. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε έτσι οι συντονιστές και οι συντονίστριες να μείνουν 5-10 λεπτά μετά τις 12.30 για να το συζητήσουμε. Μετά τις 12.30 επαναλαμβάνω. Και τώρα ο κύριος Μπουταρέλης που με τη μεγάλη υπομονή περίμενε να πει να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότηση του EDPS. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω τη δεύτερη γνωμοδότηση του EDPS για το άκουτα. Την τρίτη την εγκρίναμε για να συμπληρώσουμε εκείνη του Φεβρουαρίου του 10 όταν τα συμβαλόμενα μέρη ακόμη το συζητούσαν. Γιατί λοιπόν το κάνουμε αυτό, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες τους τελευταίους μήνες θεωρήσαμε απαραίτητο με δική μας πρωτοβουλία να κάνουμε μια δεύτερη αξιολόγηση της άκτας για να αναλύσουμε καλύτερα το τελικό κείμενο της συμφωνίας που με ιδιαίτερη έμφαση σε θέμα προστασίας ιδιωτικών δεδομένων. Αυτή η νέα γνωμοδότηση λοιπόν βασίζεται στην προηγούμενη αλλά και σε πρόσφατες υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξούν και η τελευταία υπόθεση Ντεπονιέ που είναι πολύ πρόσφατη. Κάνουμε λοιπόν μία νέα αξιολόγηση πρόσθετη και φυσικά βασιζόμαστε ιδιαίτερα στο θέμα του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων στο ψηφιακό μας περιβάλλον. Πολύ σύντομα, τέσσερα συμπεράσματα, σε τέσσερα συμπεράσματα καταλήξαμε. Πρώτον, υπάρχουν δύο ρήτρε το 27.3 και 27.4 που φαίνεται ότι ανοίγουν στην την πόρτα στην δυνατότητα λήψης μέτρων που επηρεάζουν μαζικά τη χρήση του ίντερνετ. Αυτό μας φαίνεται δυσανάλογο και παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεύτερον, πολλά από τα εθελοντικά μέτρα επιβολής, πάλι στο 27.3, θα μπορούσαν επίσης να παραβιάζουν τα προσωπικά δικαιώματα από τους προμηθευτές της πρόσβασης στο ίντερνετ πέρα από αυτά που επιτρέπονται μέχρι σήμερα. Τρίτον, δεν αρκεί νομίζουμε, δεν είναι σαφές κατά πόσον το ψηφιακό τμήμα του άκτα αφορά μόνο μαζικές παραβιάσεις προσωπικών δικαιωμάτων ή αφορά και μεμονωμένους χρήστες για μη κερδοσκοπική τους χρήση. Τελικά θεωρούμε ότι δεν έχει αρκετούς περιορισμούς και προβλέψεις όσους θα έπρεπε η άκτα. Ούτε υπάρχει καμία εγγύηση για δικαστική προστασία με με πλήρη σεβασμό της ε, αθωότητας του κατηγορουμένου μέχρι να αποδειχτεί η ενοχή του. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι ρήτρε για την επιβολή των μέτρων είναι πολύ ασαφείς και η συμφωνία είναι επίσης ασαφής ως προς τα ποια θα είναι τα μέτρα αντιμετώπισης των παραβιάσεων. για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Όπως είπα και πριν, τα είδη μέτρων που προβλέπονται στο 27.3 και 27.4 θα σήμαιναν επιτήρηση της χρήσης του Ιντερνετ από τους χρήστες για σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περίπτωση παραβίασής τους αλλά και για την πρόβλεψη της παραβίασης. Άρα απαιτείται μόνιμη επιτήρηση και εποπτεία ως προς την ανταλλαγή φακέλων όχι μόνο στα δίκτυα peer-to-peer -peer, to peer αλλα και για το κατέβασμα περιεχομένου. Αυτό μπορεί να αφορά ακόμη και ηλεκτρονικά μηνύματα. Άρα αυτή η ρήτρα για τις πιθανές παραβιάσεις θα ταυτίζονται μέσω της πληροφόρησης που κατακρατούν οι προμηθευτές πρόσβασης και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσφυγές. Και τα μέτρα θα μπορούσαν να είναι τα γνωστά, η απαγόρευση πρόσβασης κλπ. Τέτοιου είδους επιτήρηση κάτε θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό για, την, για τα προσωπικά δικαιώματα του χρήστη και το δικαίωμά του ιδιαίτερα στην εμπιστευτικότητα. Αυτό βέβαια πρέπει να θεωρηθεί να το, αυτό το λέμε αν όλα δεν γίνουν όπως υποτίθεται ότι θα γίνουν. Πρέπει να αξιολογηθεί δηλαδή το κατά πόσον τα προτινόμενα μέτρα μετά την θέση ενισχύ της άκτας είναι δυσανάλογα ή μη ως προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Πρέπει να υπάρξει μια εξισορρόπηση μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων προσωπικών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης δεν είναι σαφές ότι το ψηφιακό μέρος της άκτας θα αφορά μόνο μαζικές παραβιάσεις. Και γιατί το λέμε αυτό, γιατί το 23 ορίζει κριτήρια εμπορικής κλίμακας. Αλλά δεν είναι σαφές αν τέτοια κριτήρια θα αφορούν και τα μέτρα για το ίντερνετ. Ο ορισμός της έννοιας κριτήριο εμπορικής κλίμακας δεν είναι ικανοποιητικός. Θα προτιμούσαμε πιο σαφή αποκλεισμό από την άκτα πράξεων που γίνονται από ιδιω, ιδιώτες χρήστες για προσωπική τους χρήση. Στο 27.4 διατυπώνονται συστάσεις που ήδη υπάρχουν, αλλά προστίθενται εγγυήσει. Ιδιαίτερα σε περίπτωση προσφυγών, οπότε και ο δικαστής θα κρίνει κατά πόσον είναι δυσανάλογη ή όχι η προτινόμενη κύρωση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει παραγγελίες από τόπους εκτός της Ένωσης. Επίσης μιλήσαμε, συζητήσαμε το θέμα του εθελοντικού μηχανισμού συνεργασίας όπου οι προμηθευτές πρέπει να ελέγχουν από μόνοι τους το περιεχόμενο κάτι που ξεπερνάει κατά πολύ αυτά που επιτρέπει ο νόμος για τους προμηθευτάς πρόσβασης ο οποίος νόμος είναι σαφέστατος ως προς τα όρια της δικαιοδοσίας του προμηθευτού για θέματα καταπολέμησης ε, ε, παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος, η θεμητή ανησυχία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων είναι κάτι που το αναγνωρίζουμε καθώς και την ανάγκη για περισσότερη διεθνή συνεργασία. Αλλά υπάρχει σαφής κίνδυνος αυτή η συμφωνία, το άκτα δηλαδή ως έχει τώρα, στο μέλλον να οδηγήσει σε αλλαγή και του ίδιου του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία. Η γνωμοδότηση του, δικαστηρίου εξετάζει τη συμβατότητα με ισχύουσες συνθήκες, όχι μόνο για τον ιδιωτικό χαρακτήρα, αλλά και με πλήρη σεβασμό της, θα ήθελα να σκεφτούμε ότι εμείς το EDPS θεωρούμε πρόωρο να συμφωνήσουμε ήδη, να συνάψουμε μια διεθνή συμφωνία για αρχές που αφορούν την online εφαρμογή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όταν δεν υπάρχει καν τέτοια συμφωνία μέσα στην Ένωση. Και τα μέσα που προβλέπονται για την ενδυνάμωση του σεβασμού των, των δικαιωμάτων ε, πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι μεν θεμητά αλλά δεν είναι και από τα πιο θεμελιώδη κατ' εμάς είναι δυσανάλογο και μπορεί να βλάψει τα προσωπικά δικαιώματα γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ορισμένα θέματα, όχι από όλες τις ομάδες. Ε, θα ξεκινήσω με τον κύριο Μπουσατήλ. Ευχαριστώ πολύ Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ επίση το EDPS για την εξαιρετικά ξεκάθαρη παρουσίαση. Μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερου δύο σημεία τα οποία θέσατε. Η δυνατότητα ε, της ε, προστασίας των ISP, των προμηθευτών και η λειτουργία τους στο ίντερνετ και δεύτερον η αποτυχία της συμφωνίας να αποκλείσει κάποια άτομα που χρησιμοποιούν για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς το, στο διαδίκτυο. Ε, και η ζημία που μπορούν να προκαλέσουν. Νομίζω ότι αυτές είναι δύο ανησυχίες που θα πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά. Τώρα, το ερώτημά μου είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή η άκτα, όπως ξέρετε, είναι ένα μάλλον αόριστο κείμενο και ε, πλήρες και δεν έχει επακριβείς διατάξεις ε, και αν δούμε και αυτές τις δύο ανησυχίες ε, που αναφέραμε, γιατί να υποθέσουμε ότι οι χώρες που θα εφαρμόσουν την άκτα θα παραβιάσουν τον κοινωνικό νόμο ή παρά να θεωρήσουμε ότι θα τον εφαρμόσουν γιατί αυτού του είδους οι διατάξεις ε, το μόνο που λένε είναι ότι θα μπορούσατε να κάνετε κάτι ή θα μπορούσατε και να μην το κάνετε. Άρα λοιπόν, ε, γιατί να υποθέσουμε ότι οι χώρες μέλη θα δράσουν κατά ένα τρόπο που θα παραβιάσει το κοινοτικό δίκαιο. Γιατί υποθέτεται ότι θα κινηθούν λοιπόν κατά παραβίαση του κοινοτικού νόμου. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ρόιτεβα. Ναι, θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση και για το γεγονός ότι είχαμε την ε, δυνατότητα να ενημερωθούμε για αυτό το θέμα. Η παρουσίασή σας συμφωνεί με τις απόψεις των διαφόρων ε, ειδικών πραγματογνωμόνων που είναι γνωστές εδώ και ένα χρόνο. Και αυτή η Επιτροπή ανέλαβε ένα σημαντικό έργο. Το δικαστήριο δεν πρόκειται να ελέγξει κάποια παραβίαση. Άρα οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καθορίζονται από την προτεραιότητα του να συμπεριληφθούν στην έκθεση αυτή όλοι οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ. Και ε, όσον αφορά ορισμένους ε, κινδύνους για την παραβίαση των δικαιωμάτων πολιτών θα πρέπει επίσης να οριστούν. Έχουμε συνείδηση ότι ε, στη συμφωνία αυτή δεν υπήρχαν αυτές οι αριστείες. Αρχικά έλεγε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι χώρες μέλη διάφορα πράγματα. Αλλά επειδή διατύπωσαν κάποιες επιφυλάξεις οι πραγματογνώμονες, τελικά καταλήξαμε σε αυτού του είδους την αοριστία. Στην Τσεχία ε, μπορούν να συλλεμπευθούν ορισμένα περιεχόμενα, ενώ στη Γαλλία αντιστοίχως οι νόμοι είναι πολύ πιο αυστηροί. Άρα λοιπόν εκεί δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε αυτό το περιθώριο διαφορετικών ερμηνεών εκ μέρους των χωρών μελών. Και πραγματικά θα με ενδιαφέρει να μου πείτε κατά πόσο εσείς και οι άλλοι συνάδελφοι έχετε την άποψη ότι οι υπερασπιστές αυτής της συμφωνίας έχουν την αίσθηση ότι παρόλα αυτά θα ήταν δυνατόν εδώ και κάτω από το πρίσμα της εφαρμογής να επιληθούν αυτά τα επίμαχα προβλήματα, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω αυτή την άποψη. Αλλά ο εισηγητής θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι σημαντικό για να... και αυτό το βήμα μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Η κυρία Βέμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να πω ότι σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και για το έργο που επιτελέσατε ομολογώ ότι προσπάθησα να συμφωνήσω με την αξιολόγησή σας έχοντας κατά νου ότι δεν έχουμε επαρκή πίγνωση των ενδεχόμενων επιπτώσεων ορισμένων πτυχών αυτής της συμφωνίας. Και ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μας κάνετε μια προσεκτική ανάλυση του τι θα μπορούσε να συμβεί. Γιατί και ένα θέμα, θέμα ερμηνείας πάντοτε το τι μπορεί να συμβεί όταν εφαρμόζεται κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία. Τώρα, προσπαθώντας να κινηθούμε δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε με τον εισηγητή σε όλα τα σημεία, αλλά νομίζω ότι ορισμένα από τα θέματα που θέσετε στην εκτίμησή σας δείχνουν ότι πράγματι παραβιάζουμε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν συμφωνήσουμε με αυτή τη συμφωνία άκτα. Άρα λοιπόν είναι πολύ βοηθητική η έκθεση για μας και όχι μόνο σε σχέση με την δίσδυση στο διαδίκτυο αυτών των ε, ανθρώπων. Γιατί υπάρχει μεγάλος φόβος για, ε, για το τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες του ίντερνετ αν δεν έχουν κάποια όρια. Αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετές εγγυήσεις ενώπιον των νόμων και θυμάμαι όταν γινόντουσαν συζητήσεις στο Κοινοβούλιο για τα λεγόμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πόσο προσεκτικοί είμαστε σε σχέση με αυτές τις νομικές εγγυήσεις ε, όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ πιστική η εξολόγηση. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ. Ο εισηγητή ε, ζήτησε το λόγο εντάξει, αλλά νομίζω ότι καλύτερα να μιλήσουν όλοι και μετά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ και για την έκθεση την οποία θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη, ιδιαίτερως επειδή θέτει το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων. Αλλά όχι μόνο, δεν θέτει μόνο το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων, αλλά το ζητούμενο εδώ είναι να υπάρξουν ε, ε, να υπάρξει προστασία όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να υπάρξουν και επαρκή εφαρμοστικά μέτρα. Το γεγονό ότι αυτό δεν έχει επιτευχθεί δεν φαίνεται μόνο από την έκθεση αλλά και από προηγούμενε πραγματογνωμοσύνε που έγιναν στο πεδίο αυτό. Τώρα, έχω δύο ερωτήματα σε σχέση με την προστασία των δεδομένων. Σε ποιο βαθμό η έγκριση της άκτα θα οδηγούσε στο να υπάρξει μια επικάλυψη, μια σάφια σχέση με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την προστασία δεδομένων για τους προμηθευτές και ενδεχομένως πώς θα μπορούσαν να περιοριστούν μέσω της άκτα. Επίσης θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι οι προδιαγραφές ε, για την προστασία των δεδομένων δεν διατυπώνονται παρκώς. Θα ήθελα να μας πείτε συγκεκριμένα ποια είναι τα συγκεκριμένα πεδία, οι συγκεκριμένοι τομεί τη προστασία δεδομένων που δεν ρυθμίζονται επακριβώ μέσω τη συνθήκη, μέσω τη συμφωνία ΑΚΤΑ. Η κυρία Ένστ, ευχαριστώ πολύ το EDPS. Ε, συμμεριζόμαστε την άποψή σας ότι η συμφωνία είναι κάπως πρόημη και στη μορφή αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ε, όχι μόνο λόγω της ελληπού συνένεσης εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και πέρα από αυτό εμφανίζει πολλά προβλήματα. 12 ε, χώρες δεν, έχουν, δεν την έχουν επικυρώσει, υπάρχουν ε, τεράστιες διαμαρτυρίες κλπ. Και αν δούμε όλα αυτά θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά κατά πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο ή όχι. Εμείς ε, ως ομάδα συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας τα τέσσερα κυρίως σημεία τα οποία αναφέρεται, είναι ακριβώς αυτά τα επίμαχα σημεία που ε, θεωρούμε ότι πραγματικά είναι προβληματικά. Νομίζω ότι παραβιάζονται εδώ βασικές νομικές εγγύησεις, δεν εξασφαλίζεται η ένωμη προστασία, Εάν δούμε τι αναφέρεται σε σχέση με, την, με τις ε, δίκαιες διακδικασίες, ε, τη δίκαια δίκη, νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί αυτό μέσω της άκτα. Και τελικά πλήττονται κάποιες θεμελιώδεις ελευθερίες. Εδώ μιλούμε, αναφερόμαστε μόνο στη ζήτηση που γίνεται και που αφορά ακριβώς το μερίδιο της ΛΥΜΠΕ, της δικής μας Επιτροπής. Αλλά τι γίνεται για παράδειγμα με, τις άλλες, ε, με τα άλλα θέματα, τους άλλους τομείς, στον τομέα της υγείας για παράδειγμα. Και εδώ εγείρονται τεράστια συστήματα. Τώρα, όσον αφορά τις ε, προθεσμίες που ανέφερε ο εισηγητής, βεβαίως μπορούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες αυτές. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει από το 2010. Τελευταία φράση. Πιστεύω ότι η συμφωνία ΑΚΤΑ έχει ήδη ψηφιστεί και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις διαμαρτυρίες των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί δεν είναι δυνατόν να τις αγνοήσουμε. Και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η δική μας πολιτική ομάδα δεν βλέπει κάποια εναλλακτική δυνατότητα όσον αφορά αυτή την νομοθεσία, ακόμα και για το ζήτημα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι και ο κύριος Μαλίνοφ ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον ε, σαφή τρόπο με τον οποίο μιλήσατε. Ξέρετε, ε, ίσως από προηγούμενες συζητήσεις, ότι καταλήξαμε σε, κάποιες, σε κάποια κρίσιμα σημεία ερμηνεία του κειμένου. Θα σας ρωτήσω λοιπόν και πρέπει να απαντήσετε με ναι ή όχι. Γιατί δεν θέλω να υπάρξει πάλι κακή ερμηνεία. Είπατε ότι ό,τι κάνουν οι ιδιωτικοί χρήστες και ε, όσοι δεν έχουν ε, ε, οικονομικό όφελος ΜΕΙ ίσως θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διοξής από τους εμπλεκόμενους φορείς. Δηλαδή οι αρχές θα μπορούσαν να καταφερθούν εναντίον αυτών των ανθρώπων ΜΕΙ στο αγγλικό κείμενο. Θέλετε να σχολιάσετε, να κάνετε ερώτηση στο EDPS, θέλετε να απαντήσετε, Επιτροπή. Θα θέλαμε να έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να ε, κάνουμε μια δική μας τοποθέτηση όσον αφορά την ε, γνωμοδότηση, να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις, κυρία Πρόεδρε. Ναι, μπορείτε να κάνετε τώρα την παρέμβασή σας με σύντομες όμως ε, παρατηρήσεις και μετά θα απαντήσει και ο κύριος Μπουταρέλη συνολικά. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι και η σημερινή συζήτηση υπογραμμίζει την σημασία που έχουν ε, αυτά τα ζητήματα στην συζήτηση. <laughs> Και γι' αυτό επανειλημμένα έχουμε πει και διαστόματος του Επιτρόπου, αλλά και γενικά την σημασία τη μεγάλη που αποδίδουμε στα θέματα αυτά. Υπάρχουν μερικά πολύ σοβαρά, έχουμε κάποιες σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την γνωμοδότηση, κυρίως όσον αφορά βασική νομική τεχνική. Εν συντομία να σας μιλήσω για τα ζητήματα αυτά ο τρόπος με τον οποίο ε, φτάνει σε συμπεράσματα η γνωμοδότηση βασίζεται σε δύο ε, πεπιθήσεις. Πρώτον, ότι συστηματικά αποφεύγει αναφορά στις ε, ρήτρες διασφάλισης οι οποίες εμπεριέχονται και επίσης ρητά στο προήμιο και σε μερικά άρθρα ασχολείται με θέματα προστασίας ιδιωτικών δεδομένων και ε, αναλογικότητα. Όπως και άλλοι ε, ομιλητές ε, κατέδειξαν και ξεκινά από την παραδοχή ότι όταν θα εφαρμοστεί, δεν θα εφαρμοστεί μονάχα με τρόπο που παραβιάζει τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα παραβιάζει ταυτόχρονα και την άκτα. Ξεκινώντας από αυτή τη βάση, είναι μάλλον εύκολο να φτάσει κανείς στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πρόβλημα με τη συμφωνία. Αλλά αυτό μας εκπλήσει θα ήθελα να δώσουμε μερικά παραδείγματα και θα είμαι σύντομος. Μία από τις σαφείς παραλήψεις στην έκθεση είναι ότι πουθενά στις 60 σελίδες δεν αναφέρονται οι κύριες πρόνοιες και οι κύριες διατάξεις ε, οι οποίες αφορούν ε, τα, την προστασία προσωπικών δεδομένων, άρθρο 4 ας πούμε. Ούτε καν αυτό το άρθρο που ρητά αναφέρεται η προστασία προσωπικών δεδομένων δεν ε, αναφέρεται εδώ στην γνωμοδότηση. Επίσης, άλλο παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να εκμεύσει κατά κάποιο τρόπο το συμπέρασμα αυτό. Άρθρο 27.4. Και αν το διαβάσει κανείς εξ ολοκλήρου και όχι επιλεκτικά και κατά τμήματα, θα διαπιστώσει κανείς ότι λέει ότι ε, ε κάποιος μπορεί, μέει, σε συμφωνία με τους νόμους και τις διατάξεις Λέει δηλαδή ότι όταν και εφόσον κινηθεί κανείς με τον τρόπο που αναφέρθηκε θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον νόμο. Και δεν αναφέρει μονάχα άπαξ. Στην ίδια παράγραφο αργότερα αναφέρεται ότι αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να αποφευθεί η δημιουργία οποιονδήποτε προσκομμάτων στη... κτλ. κτλ. Και ακόμα πιο σημαντικό και οπωσδήποτε ε, σε ε, συνοχή με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς επίσης και την προστασία των ε, στοιχείων προσωπικών δεδομένων. Άρθρο 27, παράγραφος 4. Εκεί αναφέρεται τρεις φορές η προστασία των ιδιωτικών στοιχείων καθώς επίσης και η ε, συνοχή, συμβατότητα μάλλον με τους νόμους. Ε, πρόκειται λοιπόν εδώ στη γνωμοδότηση για επιλεκτική ανάγνωση. Βεβαίως ε, θα, μελετήσω με ενδελεχέστερα την γνωμοδότηση και θα ανταποκριθούμε δεόντως, αλλά εδώ έχουμε μία νομική τεχνική η οποία βασίζεται στην επιλεκτική ανάγνωση ε, της ε, συμφωνίας και η οποία, ε, και η οποία διαρκώς αποφεύγει να ασχοληθεί με συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αναφέρονται ρητά στην συμφωνία. Η κυρία Ροϊτόβα, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχω ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω γιατί με, αφού έχει υποβληθεί η συμφωνία στο Κοινοβούλιο για επικύρωση, ναι. τότε και μόνο τότε ζητήσατε να ε, εξεταστεί η συμφωνία αυτή για το κατά πόσον δηλαδή είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εμείς εδώ και δύο χρόνια αντιμετωπίζαμε προβλήματα και τώρα μόνο τη στιγμή ε, που πρέπει να επικυρώσει το Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανακάμπτει και λέει ότι θα πρέπει να εξεταστεί ε, η συμβατότητα με, το, τον νόμο της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα τι γίνεται εδώ, με ποιο τρόπο προστατεύεται ε, την ε, προστασία των ε, πνευματικών δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και καταπολεμάται την πειρατεία. Δεν καταλαβαίνω Μεγάλη σύγχυση θα δημιουργήσουμε εάν η συμφωνία εφαρμοστεί ε, και βασιζόμενη μάλιστα σε μεμονωμένες αποφάσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνούμε νομίζω οι περισσότεροι με την παρατήρησή σας. Δεν θα δώσω δυνατότητα στην Κομισιόν να απαντήσει για το θέμα αυτό γιατί ε, εμείς εδώ έχουμε εγγράψει τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της CDPS. Επομένως ε, θα πρέπει να του δώσουμε την δυνατότητα να απαντήσει για να δώσουμε μετά το λόγο και στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικέ ήταν μεταξύ τους οι περισσότερες ερωτήσεις. Γι' αυτό μπορώ να τη συνοψίσω στην απάντησή μου. Ευχαριστώ για αυτά που είπατε κύριε Μπουσουτσίλ, αλλά δεν είπα εγώ ότι η συμφωνία καθεαυτήν παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή οθεί προς την παραβίαση. Είπα επανειλημμένα και το γράφει η γνωμοδότηση ότι ανοίγει την πόρτα σε μια κατακαιρματισμένη προσέγγιση και ιδίως ανακράτος. Ως προσθέτης δραστηριότητες δεν υπάρχει ακόμη καμία συνένεση σε ενωσιακό επίπεδο για το ποιες είναι οι παράνομες δραστηριότητες. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι υπάρχουν συζητήσεις πιθανής αναθεώρησης της οδηγίας pred και εθνικά και ενωσιακά και υπάρχουν χώρες που προβλέπουν τέτοιου είδους μαζική επιτήρηση. Εμείς από ό,τι ξέρουμε είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία σαν κι αυτήν φυσικά θα περιλαμβάνει και ρήτρε όπως του άρθρου 4 που θα λένε χωρίς παραβίαση του Ευρωπαϊκού Νόμου για την προστασία των δεδομένων κτλ. Το θέμα όμως είναι πώς γίνεται αυτό στην πράξη. Πριν πάω στο EDPS είχα γράψει μια γνωμοδότηση σε εθνικό επίπεδο για τη γνωστή υπόθεση Peppermint που μοιάζει με την υπόθεση προμούζικα. Οι προμηθευτές πρόσβασης αλλά και οι διάφοροι άλλοι δικαιούχοι το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν για να εφαρμόσουν αυτή τη ρήτρα είναι να κάνουν μαζική επιτήρηση των ανταλλαγών που γίνονται μεταξύ χρηστών. Private individual for Ακόμη και για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Θα μπορούσα λοιπόν να απαντήσω λέγοντας αν οι προμηθευτές πρόσβασης από τρίτες χώρες διαμαρτυρηθούν. Τι γίνεται. Αλλά εγώ θα το θέσω αλλιώς. Πώς θα εφαρμοστεί το 27.3 και ακόμη χειρότερα το 27.4 αν δεν παραβιαστούν γνωστές αρχές διότι ένας προμηθευτής πρόσβασης υποχρεώνεται να ε, εφαρμόζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα ακόμη και ενώπιον δικαστηρίου με βάση βέβαια κάποια ισορροπία αλλά η εμπειρία δείχνει ότι πολλές περιπτώσεις και υποθέσεις προσφυγών οφείλονται σε μαζική επιτήρηση της συμπεριφοράς των χριστών. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα διατήρησης, κατακράτησης δεδομένων και επιτήρησης γιατί πολλοί προμηθευτέ κατακρατούν δεδομένα για λόγους ασφαλείας και καταπολέμησης του εγκουλήματος. Θεωρητικά λοιπόν είναι εύκολα τα πράγματα offline αλλά για τα πράγματα αλλάζουν όταν ζητάμε από έναν προμηθευτή ενώπιον δικαστηρίου να αποκαλύψει αυτά τα δεδομένα του για τους τελευταίους έξι μήνες. Πώς θα ξέρει ο δικαιούχος ο χρήστης δηλαδή αν τι ισχύει πώς θα μπορεί να ταυτίσει όλους τους υπόλοιπους. Το θέμα όμως είναι επίσης ότι αφού τα συζητάμε αυτά πρέπει να συζητήσουμε και αυτά που είπαμε όταν εγκρίθηκε η οδηγία IPRED και άλλες. Η Επιτροπή σας έχει παίξει βασικό ρόλο ζητώντας σαφείς κανόνες διαφάνειας και νομιμότητας. Επομένως το θέμα είναι γιατί ζητάμε σαφήνεια σε μερικές περιπτώσεις και όχι σε άλλες. Είστε σε θέση να δεχτείτε τέτοιου είδους ασάφεια. Το 27.3 που μιλάει για προώθηση συνεργιστικών, συνεργατικών προσπαθειών αντιμετώπιση επιτήρησης δηλαδή. Πώς θα εφαρμοστεί Μπορεί να μην υπάρχει άμεση παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά το θέμα είναι πώς νομίζετε ότι μπορούν όλα αυτά να εφαρμοστούν χωρίς παραβίαση. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Διαδικαστικό του κυρίου Πουσουτήλ. Ναι, κυρία Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τη σαφή ε, αντίθεση της Επιτροπής ε, σε αυτήν την γνωμοδότηση. Μήπως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την Επιτροπή εν ευθέτω χρόνο να μας στείλει τις, τα γραπτά της σχόλια, γιατί αυτό ε, θα έπρεπε να το έχει στη διάθεσή του ο εισηγητής μας πριν συγγράψει την γνωμοδότησή του. Συμφωνώ, ζήτησα μάλιστα και από τον κύριο Μπουταρέλη να μου πει αν έχουν λάβει γραπτά σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Καλό θα ήταν να έχουμε αναλυτικά γραπτά σχόλια έτσι ώστε να αξιολογήσουμε σωστά τα διάφορα επιχειρήματα και τα διαφορετικά μάλλον επιχειρήματα. Νεύει θετικά η Κομισιόν, άρα δέχεστε φαντάζομαι το αίτημα της Επιτροπής μας εδώ. Ωραία. Τελικές παρατηρήσεις ε, του εισηγητού και μετά θα ζητήσω να παραμείνουν δύο-τρία λεπτάκια οι συντονιστές έτσι ώστε να λύσουμε αυτό το ζήτημα του χρονοδιάγραμματος. Κύριε Δρούτσα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, κυρία Πρόεδρε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο άλλωστε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον, πρώτον ε, ε, Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ε, για τα όσα μας είπε. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω μάλιστα και για την πολύ στενή συνεργασία που είχαμε για τα θέματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να βασιστούμε στη γνωμοδότησή του. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση ε, που παρουσιάστηκε σήμερα από τον Ευρωπαίο Επόπτη είναι εξαιρετικά ε, πολύτιμη και θα μας βοηθήσει στις εργασίες της Επιτροπής μας. Καταλάβαμε από αυτά που είπατε κύριε Μπουταρέλη ότι και εσείς ενώνετε τη φωνή σας σε αυτές τις πολλές φωνές οι οποίες έχουν εκφράσει μεγάλη ανησυχία για την άκτα. Θα ήθελα όμως εγώ να αρχίσω να σκέφτομαι την επόμενη μέρα και το επόμενο βήμα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε κατανοήσει πλέον όλοι ότι η άκτα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ε, πολιτικά έχει πεθάνει, αν μου επιτρέπετε, η έκφραση. Και θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα βάλουμε στη θέση της άκτα. Και ήδη θα πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε και να συζητάμε για το τι θα ήταν καλό να έχουμε, δηλαδή ποια θα ήταν η σωστή νέα άκτα. Η συνεργασία λοιπόν με τον Ευρωπαίο Επόπτη και την ε, υπηρεσία του θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κατά αυτή την έννοια λέω. Δεν θα μπω στον πειρασμό να ζητήσω από τον επόπτη να μας πει τι θα ήταν απαραίτητο να έχουμε ε, ή τι είναι το καλό στην άκτα ή τι θα ήταν απαραίτητο να έχουμε για να έχουμε μια καλή άκτα. Ε, θα αντισταθώ όμω στον πειρασμό αυτό, θα το, συζητήσουμε μια άλλη φορά αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουταρέλη για την παρουσίασή σας. Πρόεδρος. Ξέρω ότι μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό πάρα πολύ σύντομα, αλλά καλύτερα να το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν εδώ τη συνεδρίασή μας. Επόμενη συνεδρίαση την 8η Μαΐου του 2012 στις 9 το πρωί στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, ε, συντονιστές να παραμείνουν έτσι ώστε να λύσουμε το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Οι διερμηνείς όμως είναι ελεύθεροι να φύγουν.